έλαβα από το Συμβούλιο την τοποθέτηση σε πρώτη ανάγνωση για τον κανονισμό για, το, για τη μέτρων για τα σιδηροδρομικά δίκτυα και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών δικτύων. Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θα καταγραφεί στα πρακτικά αυτής της συνόδου. Έχουμε ένα τρίμηνο στο Κοινοβούλιο για να συμφωνήσουμε στη δική μας θέση και η προθεσμία θα αρχίσει να τρέχει